το σημείο αυτό θα το ψηφίσουμε αύριο στις 12. Ε, Περνάμε στο τελευταίο σημείο. Έκθεση επίσης της ε, κυρίας Ρόβολ για την κοινή εμπορική πολιτική. Έχετε το λόγο για 4 λεπτά. Ναι. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση η οποία λέγεται και Omnibus 1 είναι προσαρμογή του εμπορικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις νέες διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας, συγκεκριμένα στο άρθρο 290 και 291. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα συναπόφασης ε, σε ζητήματα εμπορικά, κάτι το οποίο δεν έχει υπ' τη μορφή κανένα άλλο κοινοβούλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατ' ουσίαν περνάμε στην κατηγορία του Αμερικανικού Κογκρέσου και όχι στο μοντέλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μέχρι τώρα η εμπορική πολιτική κατ' ουσίαν ε, εξαιρούταν από την ε, επιτροπολογία ρητός και τον τελευταίο λόγο είχε πάντα το Συμβούλιο. Πλέον έχει τελειώσει αυτό το ειδικό καθεστώς και πλέον οι αποφάσεις όπως και σε άλλους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται από την Κομισιόν. Βεβαίως η Κομισιόν δεν το κάνει αυτό σε ένα κενό. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω σύντομα τις σημαντικότερες αλλαγές. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δούμε το Common Understanding. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με Κομισιόν και Συμβούλιο κατέληξε σε μια συνεννόηση στην οποία η εφαρμογή των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση και των εφαρμοστικών διατάξεων θα υπάγεται σε ένα ενιαίο μοντέλο. Προς μεγάλη μου κατάπληξη η Κομισιόν αυτό δεν το έλαβε υπόψη στην ε, πρότασή της, γι' αυτό η έκθεσή μου το αναφέρει και ε, προσανατολίζεται η διατύπωσή της αυτά τα οποία αναφέρονται ακριβώς σε αυτή την κοινή συνεννόηση. Δεύτερον, η εισαγωγή των πράξεων κατεξιοδότηση είναι σε όλες τις πράξεις οποίες ε, προτείνει η Κομισιόν κατόπιν η διαδικασία εξέτασης ή η λεγόμενη διαδικασία διαβούλευσης αφορά στην, ε, στις περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες έχουμε εφαρμοστικές διατάξεις. Οπότε βεβαίως αυτό θα ήταν κάτι το ιδιαίτερα μακροσκελές, γι' αυτό προτείνουμε την διαβούλευση. Κατόπιν λοιπόν η διαδικασία της ε, διαβούλευσης. Εμείς θα θέλαμε και επιβεβαιώνουμε πως αυτό πρέπει να γίνει στην πρόταση της Κομισιόν, αντί για διαβουλεύσεις οι οποίες πλέον δεν είναι απαραίτητες, κατά την ε, εισαγωγή των διαδικασιών αντι-dumping και των μέτρων κατά των επιδοτήσεων να υπάρξει υποχρέωση ενημέρωσης των κρατών μελών. Οι προθεσμίες σε αυτές τις δύο διαδικασίες δεν θέλουμε να είναι το maximum που μας δίνει ο ΠΟΕ η βιομηχανία και η εμπορικοί μας εταίροι χρειάζονται μια σιγουριά όταν προγραμματίζουν και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μικρότερες προθεσμίες. Έτσι είναι και αποτελεσματικότερα τα μέτρα. Γι' αυτό η έκθεσή μου προτείνει να μειωθούν οι προθεσμίες πλην βεβαίως κάποιων εξαιρέσεων. Κατά τα λοιπά, στους ε, περισσότερους κανονισμούς στους οποίους έχουμε τώρα, προτείνει η έκθεσή μου να έχει η Κομισιόν υποχρέωση ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κοινού. Και το πόσο σημαντικό είναι αυτό φαίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς έχουμε μία συζήτηση για την διαδικασία άκτα. διαδικασία η οποία δεν ήταν διάφανη, ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, γι' αυτό δεν μπορούμε να παρά να ενημερώνουμε συνεχώς. Η έκθεσή μου λοιπόν προσαρμόζεται σε αυτά τα οποία προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, γι' αυτό είναι αρκετά τεχνική και ταυτόχρονα είναι εξαιρετικός. Πολιτική γιατί μπαίνουμε σε μια νέα εποχή στον πάρα πολύ σημαντικό τομέα των εξωτερικών εμπορικών σχέσεων. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης τον Επίτροπο τον κύριο Ντεχούχτ. Σας παρακαλώ λοιπόν κύριε Σιόλος να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουίτσχουτ, ο Επίτροπος Σιόλος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτρέψτε μου εξ αρχής να πω ότι Επίτροπος Ντεχούχτ είχε ήδη σχεδιάσει ταξίδι στο εξωτερικό σήμερα και λόγω του ότι το σημείο προσθέθηκε την τελευταία στιγμή στην ημερήσια διαταξή δεν ήταν δυνατό να τροποποιήσει το ταξίδι του όπως ε, θα ήθελε άλλωστε για να είναι και σήμερα απόψε εδώ μαζί σας. Γι' αυτό μου ζήτησε να μιλήσω εκ μέρους της Κομισιόν Προθέματος. Είμαστε ευγνώμονες προς την κυρία Κίστχουτ Ρόβολ και τον σχετική τον κύριο Μωρέιρα καθώς και στα άλλα μέλη της ΣΥΝΤΑ για την επικοδομητική προσέγγιση στην πρόταση αυτή. Σημαντική πρόταση καθώς είναι το πρώτο βήμα για να ευθυγραμμιστούμε με το νέο καθεστώς όσον αφορά τις κατεξουδότησης πράξεις. Θέλουμε βεβαίως της κοινή εμπορικής πολιτικής. Η Κομισιόν δεσμεύεται να συνεχίσει να συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε ο φάκελος να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Αυτή την εβδομάδα έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό τροπολογιών. Βεβαίω είναι αδύνατο να τις σχολιάσω όλε μία προς μία. Πρόκειται για εργασία που θα διεκπαιρεώσουν τα τρία θεσμικά όργανα. Περιορίζομαι σε μερικές γενικές παρατηρήσεις. Καταρχήν και καταρχάς η Κομισιόν μπορεί να δεχθεί όλες τις τροπολογίες που προτείνουν τη συμβουλευτική διαδικασία, τις διαβουλεύσεις για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων. Γνωρίζουμε ότι η κατεξουδότηση πράξης πρέπει να αποτελέσουν και έναν μηχανισμό διασφάλιση εναντί της Κίνας. Τρίτον, η Κομισιόν ευχαριστεί για τις τροπολογίες που αφορούν τον κανονισμό anti-dumping. Υποστηρίζουμε το πνεύμα των τροπολογιών επίσης που αφορούν το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή νέων κανόνων επιτροπολογίας στο πλαίσιο της νομοθεσίας αντι-dumping. Παρ' όλα αυτά, οι τροπολογίες αυτές δημιουργούν ορισμένα πρακτικά προβλήματα, άλλες φορές νομικά προβλήματα. Η Κομισιόν ελπίζει ότι θα βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος να λύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο της συζήτησης που θα γίνει μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων μετά από την ψηφορία στο Κοινοβούλιο. Κλείνω λέγοντας ότι η Κομισιόν εκτιμά βαθύτατα την εργασία σας ως τώρα. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ώστε σε το χρόνο να κλείσουμε τον φάκελο αυτό. Πρόεδρε, με την ευκαιρία αυτή, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. παίρναμε στους εκπροσώπους των ομάδων και το ΕΛΚ, ο κύριος Κασπαρή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, λυπούμε ιδιαίτερα για το ότι συζήτηση για αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα γίνεται αργά το βράδυ, χωρίς ε, παρουσία κοινού και του αρμοδίου επιτρόπου. Γιατί δεν θέλω να κατηγορήσω τον κύριο Επίτροπο. Απλά λυπούμε για το ότι αυτή η έκθεση η οποία αναφέρει και ορίζει πάρα πολλά πράγματα για τα οποία πάλευσε την τελευταία δεκαετία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έκθεση αυτή λοιπόν ε, δεν ε, ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο ε, φαίνεται στην δημοσιότητα. Γιατί, γιατί αυτό το οποίο έκανε η κυρία Ρόβολ και οι σκιώδες ηγητές ορίζει πάρα πολλά πράγματα και ε, αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί από το Δεκέμβριο του 2009 και τώρα με τον κανονισμό αυτό ε, έχουμε αρμοδιότητες οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στον κόσμο. Ίσως πράγματι όπως αναφέρατε να είναι συγκρίσιμη η κατάσταση στη ΣΥΠΑ, αλλά αν δείτε άλλα κοινοβούλια, π.χ. τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή δεν είχε ποτέ τέτοιες αρμοδιότητες όσον αφορά την εξωτερική εμπορική πολιτική αυτά τα οποία έχει λέει τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ λοιπόν τους ε, συναδέλφους, ε, ειδικά όσον αφορά τα μέσα ε, κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων. Ήταν κάτι το οποίο χρειαζόμασταν επιγόντως. Ευχαριστώ ιδιαίτερα επίσης τους συναδέλφους για το ότι κινήθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια στον τομέα αυτών και θα ήθελα επίσης να πω πως θα επιθυμούσα ειδικά στον τομέα της ε, εμπορικής πολιτικής να συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη την οποία φέρουμε. Δεν είμαστε μόνο άνθρωποι οι οποίοι θα φωνασκούμε και δεν τους παίρναν σοβαρά όπως γινόταν πριν το 2009 αλλά πλέον θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε έχω ακόμη μια παρατήρηση την οποία θα ήθελα να κάνω εδώ πέρα θα πρέπει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο έτσι ώστε και η διοίκηση του Κοινοβουλίου να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να ελέγχει την όλη διαδικασία που λέγαμε επιτροπολογία. Σας ευχαριστούμε κύριε Κάσπαρη, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες 1,5 λεπτό ο κύριος Μορέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι πέρασε πολύ καιρό από όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξετάσει την κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης και τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις κατεξουσδότηση πράξεις και τις εφαρμοστικές πράξεις που είναι αποτέλεσμα ε, της συνθήκης Λισαβόνας. Θυμηθούμε τι λέει η Λισαβόνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έχει νομοθετική εξουσία μόνο κατόπιν κατεξουσδότηση πράξεων που υπόκεινται στον έλεγχο και υποπτία των δύο αρχών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δεύτερον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι το Συμβούλιο ε, θα πρέπει να υπόκειται στον έλεγχο των κρατών μελών. Στα πλαίσια του εμπορίου και της εμπορικής πολιτικής είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης και όχι των κρατών μελών. Και η πολιτική θα πρέπει να ακολουθεί την κοινοτική μέθοδο πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγκριση από τα δύο άλλα θεσμικά όργανα και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί όσον αφορά την εφαρμογή νέων μέτρων που απορρέουν τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο όλων των νομοθετικών εκρών της ενώσεως αλλά θα πρέπει να θεωρήσουμε ως κατεξουσιοδότηση πράξη όλες τις υποθέσεις εκείνες κατά τις οποίες καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει νομοθετικές πράξεις. Δεύτερον, όσον αφορά τις εφαρμοστικές διατάξεις, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να έχουν δικαίωμα βέτο όσον αφορά τι εκτελεστικέ εξουσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι είναι αποκλειστικό θέμα η εμπορική πολιτική τη Ένωση. Εάν είχαν δυνατότητα αρνησικυρία στα κράτη-μέλη, αυτό θα έπρεπε να προβλέπεται μόνο σε εξαιρετικέ περιστάσει και δεν θα πρέπει να είναι κανόνα. Τέλο, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Βαρχόλ, για την έξοχη δουλειά που έκανε και για το πνεύμα το συμβαστικό που ακολουθήθηκε σε όλη τη διαδικασία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Για του Δημοκράτε Φιλελευθέρου, για 1,5 λεπτό, η κυρία Κοχμέριν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Από τη συνθήκη τη Λισαβόνα το, έχουν αλλάξει τα πάντα στην ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Υπάρχει μια τελείως νέα νομική βάση και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπετε τα αποτελέσματα της νέας συνθήκης. Στο θέμα αυτό, το οποίο συζητάμε τώρα, ε, τα ζητήματα είναι μόνο εκ πρώτης όψεως ε, τεχνικά. Όσον αφορά δηλαδή τις ε, εφαρμοστικές διατάξεις και τις πράξεις ε, κατευσιοδότηση αλλά και τα δύο αυτά κρύβουν πολύ συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα. Σκεφτείτε μόνο τις προθεσμίες στα μέτρα anti-dumping ή τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων. Εδώ πέρα ο χρόνος κατά κυριολεξία είναι χρήμα. Και οι νέε απαιτήσει διαφάνειας για μη εμπιστευτικέ πληροφορίε, είναι πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσες για το κοινό. Ανέφερε η κυρία Ρόβολτ ε, τη ΑΚΤΑ. Εάν είχαμε μια ανάλογη διαφάνεια από την αρχή στο θέμα αυτό, ποιο ξέρει θα ήταν τελείως διαφορετική η συζήτηση αυτή, ίσως να μην είχε γίνει τόσο έντονα. Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή θα πρέπει βεβαίως απλά να ευχαριστήσουμε την ε, η συγγήτρια η οποία με σταθερό χέρι καθοδήγησε την όλη αυτή η υπόθεση και νομίζω πως ε, και εδώ πέρα γρήγορα θα οδηγηθούμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ κυρία Κοχμερίν και περνάμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Δύο λεπτά η κυρία Κέστιγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η έκθεση αυτή για την κοινή εμπορική πολιτική ε, η οποία βεβαίω είναι πιο γνωστή υπό το όνομα Omnibus 1 είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εμπορική πολιτική. Δεν θα πρέπει να μας ξεγελάει το τεχνικό ζήτημα και η πολυπλοκότητα. Έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα μπροστά μας. Ορίζει την Επιτροπή Εμπορικών ε, ζητημάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ε, συνομιλητή σε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Ήδη αναφέρθηκε η άκτα. Θα ήθελα να αφαιρθώ εγώ σε τρία σημεία τα οποία κατά την αποψή μου πρέπει να τονίσουμε γιατί έχουν μεγάλη σημασία. Πρώτον, η διαδικασία εξέτασης. Η διαδικασία εξέτασης, ναι, αλλά πρέπει εδώ πέρα πάντα να υπάρχει η δυνατότητα να βλέπουμε τα μέτρα τα οποία απαιτούνται να ληφθούν σε καταστάσεις έκτακτες και ε, οξυμένες. Δεύτερον, το εύρος της διαδικασίας διαβούλευσης ε, η στενή συνεργασία των ενδιαφερομένων και των θεσμικών οργάνων εξακολουθεί να είναι αναγκαία. Τυχόν παρεξηγήσεις μπορούν έτσι να αναγνωριστούν πολύ πιο γρήγορα και να ληφθούν υπόψη στις αποφάσεις. Τρίτον, οι προθεσμίες, ε, μια γρήγορη επίλυση των ζητημάτων προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων, το να γίνουν πιο σύντομες οι προθεσμίες ωφελεί και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στους εμπορικούς εταίρους και μπορούν να ανακλητώσουμε δύο μήνες σε όλη αυτή την υπόθεση. Θα πρέπει λοιπόν βεβαίως να φροντίσουμε να ολοκληρώνουμε γρηγορότερα τις υποθέσεις. Χαιρετίζω λοιπόν την έκθεση και ευχαριστώ ακόμη μια φορά την εισηγήτρια για την εξαιρετική της εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κέστιγκερ. Για ένα λεπτό ο κύριος Γιώργ Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Εισηγήτρια. Θεωρώ πως μπορούμε να πούμε το εξή. Η Ευρωπαϊκή εξωτερική εμπορική πολιτική ήταν πάντα κάτι στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε να επιδείξει μεγάλες επιτυχίες. Γιατί, Γιατί είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνεται στοχευμένα. Και τώρα με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε την εξή κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά είναι πλέον ισότιμος συνομοθέτης στο σύνολο αυτής της διαδικασίας και υποθέτω πως με βάση αυτά τα γεγονότα η πολιτική αυτή θα είναι ακόμη πιο επιτυχής βεβαίως. Είναι κάτι το πολύ πολύπλοκο όλες αυτές ε, οι διαδικασίες να ενταχθούν στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Θεωρώ όμως πως ε, με το Omnibus 2 και με την συνεργασία της ηγητρίας καταφέραμε να βρούμε ένα σύστημα στο οποίο αφενός ε, το οποίο εμείς εμπιστευόμαστε αλλά υπάρχει βεβαίως και έλεγχος και η Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να δράσει όπως ε, θεωρεί ότι πρέπει να δράσει και αυτό, γιατί αυτό το οποίο συνέβη με την άκτα ελπίζω ότι δεν θα επαναληφθεί ξανά. Σας ευχαριστούμε και ελάχιστη περνάμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye. Ποιος... Μόνο η κυρία Μπασέσκου έχει ζητήσει λοιπόν το λόγο. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, υποστηρίζω την τροποποίηση των 26 πράξεων του Κοινοβουλίου που αφορούν την εμπορική πολιτική για να ευθυραμιστούμε με το νέο σύστημα των κατεξουδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων. Έτσι ενισχύεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί στον τομέα τη κοινή εμπορική πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη θα είναι πιο ανταγωνιστική στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε πρωτοβουλίε για να λάβει του ρόλου και τα καθήκοντα που του αναλογούν μετά από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση τη Κομισιόν να προβαίνουμε στην ε, διαδικασία εξέτασης, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Τα μέτρα διασφάλισης είναι πολύ σημαντικά εμπροκειμένου και όντως σωστό είναι να δούμε σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητα. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπος. Πρόεδρε, κάποιες τελικέ τελικές παρατηρήσεις. Όπως έδειξε και η συζήτηση, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι τεχνικά εξαιρετικά πολύπλοκο όμως αφορά και πολλά σημαντικά νομικά κείμενα στον τομέα της εμπορικής πολιτικής. Δικαιολογείται λοιπόν ο χρόνος που αφιερώσαμε για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα το συντομότερο δυνατόν. Κατά δεύτερο λόγο, η Κομισιόν εκφράζει την ικανοποίησή της για τις τροπολογίες εν γέννη του Κοινοβουλίου και θα έχει τη χαρά να συνεργαστεί για τη συζήτηση στα πλαίσια του τριμερός διαλόγου. Τέλος, το θεμελιώδες ζήτημα παραμένει. Με ποιο τρόπο θα διαχειριστούμε από εδώ και πέρα τα μέσα που διαθέτουμε για να υπερμηνθούμε της εμπορικής μας πολιτικής. Αυτά θα τα κρίνουμε κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου. Ευχαριστούμε θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εισβάθος εργασία του επί του θέματος και σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Επίτροπος θα είναι στο πλευρό σας για να καταλήξουμε στα θέματα εμπορικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ Επίτροπε. Η κυρία Κουιστχούτ Ρόλ. Ναι, σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κοιόδης εισηγητές και ευχαριστώ κύριε Σιόλος την Επιτροπή η οποία επέδειξε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με διαβεβαίωση και για αυτήν στο μέλλον. Αύριο θα ψηφίσουμε όλες τις ε, τροπολογίες και θα έχουμε και τελική ψηφοφορία. Στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα θα ήθελα να έχω και τη στήριξη της Ολομέλειας στο θέμα αυτό. Μόνο έτσι μπορώ με τους συναδελφούς μου να πάω σε ένα τριμερή διάλογο. Ελπίζω να τελειώσουμε σύντομα γιατί όλοι θέλουμε ε, να συμβιβαστούμε. Το θέμα μας εδώ πέρα είναι η ουσία. Δηλαδή να ε, προσαρμοστούμε στο νέο νομοθετικό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συνεργασία και καλή σας νύχτα. Υποθέτω πως όλοι για ύπνο θα πάμε. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, ευχές. Θα ψηφίσουμε αύριο, θυμίζω, στις 12.